przewodniczący! E, koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάμε την συνεδρίαση. Έχετε λάβει τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Υπάρχουν παρατηρήσεις ή ενστάσεις όχι. Και ως εκ τούτου εγκρίνονται τα πρακτικά στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Προβλέπεται δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χρηματοπιστική διακυβέρνηση, την οικονομική διακυβέρνηση, την Ευρωζώνη, την εποπτεία των εθνικών προϋπολογισμών. Κύριε Παρόσο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές. Η οικονομική διακυβέρνηση αποτελεί κρίσιμο η πρόκληση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ο πρόεδρος Ντελόρ είχε εκθέσει την ανάγκη για ένα συντονισμό ενισχυμένο των οικονομικών πολιτικών. Ήδη το 1993 πολλά κράτη-μέλη είχαν απορρίψει την πρόταση αυτή. Όταν η πρώτη επιτροπή της οποίας είχα την τιμή να ηγηθώ, επανέφερε το θέμα αυτό με την έκθεσή μας για τη δέκατη επέτειο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης του 2008 πάλι δεν μας άκουσαν πολύ. Πριν όμως εγώ επέμεινα να δοθεί κατάλληλη απάντηση στο ζήτημα της οικονομικής διακυβέρνησης και στις κατευθυντήριες γραμμές για την τρέχουσα θητεία μας, τις οποίες και συζητήσαμε περίπου πριν από ένα χρόνο. Ο Επίτροπος Ρέν, εδώ παρόν, με τη σειρά του συζήτησε κατά την ακρόασή του με τους βουλευτές το θέμα αυτό και ήδη τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταθέσει την πρόθεσή της για υποβολή προτάσεων για την ενίσχυση οικονομικής δικυβέρνησης Ευρώπης και ιδιαίτερα στη ζώνη του ευρώ. Η κρίση μας δικαίωσε δυστυχώς. Όμως πλέον έχει αναγνωριστεί ότι είναι κατεπίγουσα ανάγκη ανάδειξη αυτής της συζήτηση και τώρα υπάρχουν οι συνθήκε εκείνε που μα επιτρέπουν να προχωρήσουμε ως πραγματική οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Και έτσι στι 12 Μαου κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτάσει τη, οι οποίε τροφοδοτούν τη συζήτηση, το διάλογο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερω στι εργασίε τη Task Force, τη οποία ηγείται ο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Επιτροπή εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή τη για την πρόοδο των εργασιών αυτών και, και για τη συνένεση που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, η οποία και εκδηλώθηκε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προκειμένου να διαφυλαχθεί αυτή η δυναμική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη Τετάρτη υιοθέτησε επιπλέον ένα σύνολο προτάσεων που μπορούν να μεταφραστούν σε νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία στη συνέχεια θα μα επιτρέψει, εν ευθέτω χρόνο, να προχωρήσουμε σε υλοποίηση των μέτρων αυτών το 2011 ήδη. Οι προτάσει αυτέ ακολουθούν μία πάγια γραμμή, ότι πρέπει δηλαδή να δράσουμε υπό το νομικό καθεστώ που έχουμε αυτή τη στιγμή. Φυσικά, οι πολίτε, που μας προσφέρει η συνθήκη απαιτούν Λισαβόνας πρέπει και οφείλουν να αναπτυχθούν πλήρως, να αξιοποιηθούν πλήρως. Δεν έχουμε πλέον χρόνο να περιμένουμε. Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, η οικονομία απαιτούν νεε πρωτοβουλιε Και πρέπει να αποφασίσουμε και να δράσουμε εμέσω. Στα αγγλικά. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, εξότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Η οικονομική κρίση μα έχει θέσει ενώπιον ε, μια σειρά πολύ σημαντικών δοκιμασιών και το ζήτημα τη οικονομική διακυβέρνηση είναι μόνο μία πτυχή τη ανταπόκριση που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κρίση. Η ανταπόκριση έχει και άλλε διαστάσει και συνεπάγεται και μια άρδιν μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και μια εποπτική αρχιτεκτονική σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω είπα σήμερα το πρωί, μπορούμε τι επόμενε ημέρε να προσβλέπουμε σε μια συμφωνία και παρακαλώ όλε τι πλευρέ να διαφυλάξουν την ε, ε, ένταση των συνομιλιών έτσι ώστε να προχωρήσουμε το χύτερο δυνατό και να προχωρήσουμε στην ε, υλοποίηση και των δεσμεύσεων μας επίπεδο της ομάδας των 20 G20 στα θέματα αυτά. Η οικονομική σταθερότητα και με το πρόγραμμα για την Ελλάδα και με τους μηχανισμούς για το ευρώ συνολικά αλλά και για το πρόγραμμα ανάπτυξη για θέσεις εργασίας εγγράφονται στη στρατηγική του 2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανταπόκρισή μας στην κρίση είναι ολιστικού χαρακτήρα. Σταθεροποιούμε, ε, παγιώνουμε και εξυγχρονίζουμε και προετοιμάζουμε ταυτόχρονα την οικονομία της αγοράς μας για να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μερόν για τους πολίτες μας. Επιτρέψτε όμως τώρα να επικεντρωθώ στην διακυβέρνηση. Η πρόκληση των τελευταίων μηνών επικεντρώνεται στο κατά πόσον μπορούμε να ανταποκριθούμε στι πιέσει με συνθήκε οικονομική και νομισματική σταθερότητα. Έχουμε μέτρα, έχουμε θεσμού που μπορούν να μα επιτρέψουν να αντιδράσουμε. Ε, έχουμε πραγματικού κινδύνου αντιμετωπίσει. Έχουμε επιτυχώ ε, σταθεί όρθια απέναντι σε αυτού του κινδύνου και τώρα προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα μηχανισμό που θα μα επιτρέπει να προλαμβάνουμε τέτοιου κινδύνου. Και γι' αυτό θα ήθελα να υποβάλω στο Κοινοβούλιο τις ιδέες που έχει καταγράψει με την έκθεσή της του 10 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι οποίε επανέλαβε και με την ανακοίνωση της 20 Ιουνίου. Προχωρούμε τώρα στην επόμενη φάση με τις επτά νομοθετικές προτάσεις που σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει στις αρχές Σεπτεμβρίου, το ταχύτερο δυνατό δηλαδή. Και Προσβλέπουμε στη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα από τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπό την Task Force βεβαίω, ε, τη οποία ηγείται ο πρόεδρο του Συμβουλίου, αλλά και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε οι προσπάθειε να είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εντατικέ, με συνθήκε συνεργασία, συνδιαλλαγή και ταχύτατη υιοθέτηση των προστάσεων. Η οικονομική διακυβέρνηση σημαίνει κανόνε συνολικού, ε, γενικού και αποτελεσματικού Έχουμε περιθώριο ευρύτατο που προσφέρει η νομική βάση η συνθήκη για να προχωρήσουμε τέτοια μέτρα και όπως είπα μας δίνει τις κατάλληλες απαντήσεις. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρότερο καθεστώς εποπτείας, αυστηρότερο δηλαδή αλλά και ευρύτερο, που θα καλύπτει και τους προϋπολογισμούς, τα δημοσιονομικά δηλαδή μέτρα, ε, και τη μακροοικονομική αλλά και τη διαρθρωτική πολιτική. Και έτσι κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, ταυτόχρονα όμως έχουμε και την αλληλεξάρτηση του ενός από τον άλλον που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της οικονομίας μα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα, ότι χρειάζεται περισσότερο συντονισμό και εδώ κέριο στοιχείο είναι η ευρωπαϊκή αρχή με τα, με τα με το σύστημα των εξαμήνων, την παρακολούθηση δηλαδή των προγραμμάτων, των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμιση ταυτόχρονα που θα μας επιτρέπει να έχουμε μια κοινή προσέγγιση. Αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική θα αποτελεί κέρδος και για τα κράτη-μέλη, καθώς αυτά θα προχωρούν στην συζήτηση, του προγραμματισμού και την έγκριση των εθνικών του προπολογισμών με βάση εθνικέ διατάξει. Δεύτερον, χρειάζεται η αξιοπιστία που συνεπάγεται η καλύτερη υλοποίηση των μέτρων, δηλαδή προσδιορισμένες, τόσο, προσδιορισμένα τόσο κίνητρα όσο και κυρώσεις, ως, ένα, ως μια εργαλειοθήκη η οποία θα βοηθήσει προληπτικά και κατασταλτικά στην επιτεύξη των στόχων. Και έτσι θα προσδιορίζονται και τα κριτήρια των ελλημάτων, αλλά και του χρέους. Τα πιο αυστηρά μέτρα βεβαίως θα είναι αυτά τα οποία θα ελπίσουμε ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε. Θα είναι τα μέτρα εκείνα τα οποία θα αποτελέσουν το κίνητρο για συμμόρφωση στους κανόνες. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι οι κανόνες θα πρέπει να είναι αρκετά στεναροί, αρκετά αυστηροί για να προκαλέσουν τη συμμόρφωση. Αυτό, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν σημαίνει ότι ε, το να έχουμε ένα πολύ χαλαρό σύστημα μπορεί να ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμφωνούν και να τηρούν τους κοινού αυτούς κανόνες. Και έτσι οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπον ώστε να ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη ισοδύναμα, σε ισότιμη βάση. Το Δακοινοβούλιο, το σας διαβεβαιώνω, ότι ασφαλώς και αυτό θα πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να είστε ήσυχοι ότι αυτό είναι το καθήκον μας. Επίσης, οι κυρώσει έχουν να κάνουν, προβλέπεται ότι θα αναπτυχθούν από ένα ολόκληρο δυναμικό μέτρο από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, ε, δηλαδή τα κράτη-μέλη τα οποία επανειλημμένως δεν τηρούν τους δημοσιονομικούς κανόνες θα χάνουν τη χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και μάλιστα αυτός ο κανόνας θα είναι σχεδόν αυτοματοποιημένος όπως ε, επί με το διορθωτικό μέτρο της σταθερότητας ε, του Συμφώνου σταθερότητα. Δεν πρέπει να περιμένουμε δηλαδή να αναπτυχθεί η κρίση μέχρι να, πριν να, κατα, να επιβάλλουμε τα μέτρα. Πρέπει να επιβάλλουμε τα μέτρα το ταχύτερο δυνατό τόσο σε επίπεδο κινήτρων όσο και σε επίπεδο κυρώσεων. Προληπτικά βέβαια είναι καλύτερο να δράσουμε από ότι κατασταλτικά αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γνωρίσουμε ότι θα χρειαστεί η κατασταλτική δράση σε ορισμένες περιπτώσεις. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί για να ε, προσέξουμε την συμπεριφορά των κρατών και τον προπολογισμό του στι λεγόμενε περιόδους των παχαίων αγελάδων. Αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και επίση θα υπογραμμίσω ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην δημοσιονομική ε, πολιτική. Τέτοιου είδου προοπτικέ δεν επαρκούν. Πρέπει να έχουμε τα μέσα να διαπιστώσουμε και τι μακροοικονομικέ ανισορροπίε οι ανισότητε μέσα στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα δε για, τον, για, τον, ε, για το ζώνη του ευρώ. Θα έχουμε λοιπόν επαρκή αριθμό δικτών που θα μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε τις ανισότητες, τις ανισορροπίες και να προτείνουμε μέτρα. Αυτό πάλι απαιτεί συγκεκριμένους μηχανισμούς επιβολής των μέτρων αυτών και λειτουργία των μηχανισμών. Αυστηρία λοιπόν δημοσιονομικά μέτρα και ταυτόχρονα μεταρρυθμίσεις, καινοτομία, νεοτερισμός, ανάπτυξη και νέε θέσει εργασία για το μέλλον. Αυτά είναι άλλωστε και το περιεχόμενο τη στρατηγική μα για το 2020. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από δύο εβδομάδε περίπου υιοθέτησε αυτή τη στρατηγική και τώρα μένει να την υλοποιήσουμε έτσι ώστε οι ευρωπαϊκέ και οι εθνικέ πολιτικέ να είναι ευθυγραμμισμένε για την ανάπτυξη του, ε, του αέναου εκείνου και θετικού κύκλου που θα μα επιτρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον επιτυχώς. Πέμπτον, επιτρέψτε μου να φερθώ τώρα στην ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών για να παρακαλέσω του πάντε να προχωρήσουν ταχύτερη δυνατή υιοθέτηση των σχετικών μέτρων. Θα θέλω να υπογραμμίσω την ιστορική διάσταση των μέτρων που καταθέτουμε, που αποτελούν μια, πρόκληση, μια απάντηση στι προκλήσει τι οποίε αντιμετωπίζει το ενιαίο νόμισμα στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα όμω θα έχουν και σημαντικό αντίκτυπο και στι παγκόσμιε χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Είναι η ώρα να δώσουμε πλέον στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση τα εργαλεία που χρειάζεται για να μπορέσει να τιμήσει την εντολή τη και να εξασφαλίσει τη σταθερότητά τη. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν. Έχουμε να κάνουμε με το μέλλον το ίδιο του ευρώ, έχουμε να κάνουμε με το μέλλον, θα μπορούσα να πω ακόμη, του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Άρα θα πρέπει να αποδείξουμε χωρίς την παραμικρή εμφολία ότι έχει αλλάξει η κατάσταση και ότι η χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση την οποία εμείς προτείνουμε είναι ριζοσπαστική, είναι κάτι το καινούριο. Σταθερότητα, προοπτικές, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση είναι το νέο σύστημα που προτείνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι και με την επιτήρηση των προπολογισμών και τα ερωτικά ταμεία μπορούμε να προχωρήσουμε στη στρατηγική που θέλουμε για την Ευρώπη του 2020, που είναι μια στρατηγική ενιαία και όχι ένα συνονθήλευμα διαφορετικών στρατηγικών. Είναι μια και μόνη στρατηγική για όλη την Ευρώπη, η οποία όμως μπορεί να υπάρχει μόνο εφόσον υπάρχει ένα ενιαίο οικονομικό σύστημα διακυβέρνηση. Το σύστημα των κινήτρων και των ε, όμως ωστόσο, θα πρέπει να υπαχθεί στην ευθύνη των κρατών μελών, τα οποία έχουν υιοθετήσει ήδη το ενιαίο νόμισμα και ω εκ τούτου έχουν συμμορφωθεί σε αυτό το ε, νομικό πλαίσιο. Έχουν ένα κοινό αγαθό να μοιραστούν τα κράτη-μέλη και είναι το ευρώ. Δεν μπορεί λοιπόν η συμπεριφορά κάποιων κρατών μελών να θέτει σε κίνδυνο τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, το αγαθό το οποίο ανήκει και στα άλλα κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν ζήτημα και συνοχή τη Ευρωπαϊκή Έννοια και συνέπεια έναντι τη Ευρωπαϊκή Έννοια. Ενώ ταυτόχρονα φυσικά διαφυλάσσονται και οι ιδιαιτερότητε των κρατών μελών τη ε, ζώνη του ευρώ, αλλά και ο σεβασμό εκείνων των οποίων δεν είναι μέλη τη ζώνη του ευρώ. Χρειάζεται φιλοδεξία, χρειάζεται θάρρος, παρησία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει σαφές μήνυμα σε όλους, σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι μπορούμε να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Τα τρία θεσμικά όργανα εργαζόμαστε από κοινού, με συνέπεια και σε πνεύμα αγαστή συνεργασίας για να αναπτύξουμε καλούς κανόνες, μέτρα και συστήματα για το μέλλον το κοινό μας μέλλον, το κοινό της Ευρώπης και είναι απαραίτητο οι εταίροι σε ολόκληρο τον κόσμο να αντιληφθούν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ότι θα μετέλθουμε για οδήποτε πρόσφορο μέσο για να φυλάξουμε την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως καθήκον να διαφυλάξει τη ε, συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της και θα κάνει κάθε τι έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. ευχαριστώ για την προσοχή σας. Dziękuję, e, panie przewodniczący za ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που παρουσιάσατε τη συζήτηση και το θέμα και τώρα να δώσω το λόγο στους ε, εκπροσώπους ε, των ε, πολιτικών κομμάτων. Πρώτα απ' όλα, κύριε Μορφανκόλ, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πολύ σημαντική ε, η ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ε, οικονομικής διακυβέρνησης. Δεν πρέπει να περιμένουμε την, ε, την ολοκλήρωση των εργασιών της Tax Force του Συμβουλίου. Εμείς στο ΕΛΚ Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι προσπάθειες, ούτω ώστε ε, να υπάρξει μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση. Θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική συνεργασία για να προωθήσουμε την κοινοτική μέθοδο. Δεν θα δημιουργήσουμε νέα θεσμικά όργανα, αλλά θα δώσουμε τη δυνατότητα ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει έναν εξάρτητο και δυναμικό ρόλο. Το Συμβούλιο θα πρέπει να ε, εξασφαλίσει ένα δημοκρατικό έλεγχο, να προωθήσει μάλλον το δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά συστατικά για την ε, επιτυχή εφαρμογή των προτάσεων που θα μας παρουσιάσετε το Σεπτέμβριο. Ε, τα εθνικά προγράμματα, οι μεταρρυθμίσεις, ε, τα δύσκολα μέτρα που θα ληφθούν στα διάφορα κράτη-μέλη είναι απαραίτητα για να υπερασπιστούμε την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών και των οικονομιών μας. Και με αυτόν τον τρόπο ε, νομίζω θα πείσουμε και τους Ευρωπαίους πολίτες. Περιμένουμε πολλά από το ενισχυμένο και μεταρρυθμισμένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Επίσης, ε, τα κίνητρα και οι κυρώσεις είναι πολύ σημαντικές ε, που προβλέπονται. Όλα αυτά βεβαίως θα εξαρτηθούν, ε, η αποτελεσματικότητά τους θα εξαρτηθεί από το σεβασμό από τους διάφορους εμπλεκόμενους. Η ομάδα του ποδοσφαίρου των της χώρας μου είπε ότι το θέμα δεν είναι να μιλάμε, αλλά να δρούμε, να παίζουμε. Ε, λοιπόν, πρέπει να περάσουμε στην πραγματική εφαρμογή της ε, οικονομικής διακυβέρνησης. Δεν πρέπει να μιλάμε απλώς, αλλά να δρούμε. Ε, είναι σημαντικό επίσης και η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων. Το Συμβούλιο ασχολήθηκε με την έκθεση de la Τώρα είναι και καινή ώρα να πέρασουμε στη δράση. Σε δράση νομοθετική, σε εποπτεία των ε, ιδρυμάτων αυτών όλα θα ξεκινήσουν από την 1η Πρώτου 2011. Όλα εξαρτώνται από το πώς θα αντιδράσει το Συμβούλιο. Θα πρέπει ε, αυτό το μήνα στο ΕΚΟΦΗ να υπάρξει συμφωνία όπου μαζί με τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμφωνήσουμε για τον ε, έλεγχο και για την χρηματοπιστωτική εποπτεία. Το Κοινοβούλιο όμω θα προσπίσει τα συμφέροντά του. Όχι μόνο για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μα, αλλά για να υπερασπιστούμε του ε, πολίτε μα που μα εξέλιξαν, τη σταθερότητα των χρηματαγορών, ούτω ώστε να ατενίσουμε το μέλλον με εμπιστοσύνη. Πρόεδρος. Τώρα, από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, το λόγο έχει ο κύριος Χιούγκς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Παρόζο και κύριε Ρεν, βλέπουμε ότι οι προτάσει σα ε, ε, στερούνται ισορροπία. Αυτή η πρόταση δεν μπορεί να εξεταστεί απομονωμένα από το θέμα τη ανάπτυξη και τη απασχόληση. Ε, τα ε, περαιτέρω μέτρα λιτότητα θα οδηγήσουν σε μια ε, συνεχιζόμενη περίοδο μείωσης της ανάπτυξης, της απασχόλησης, μείωση απασχόλησης και αύξηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν νομίζω να πιστεύετε ότι πρέπει να πληρώσουμε αυτό το τίμημα για να πετύχουμε τη φορολογική εξυγίανση και όμως ακολουθείτε το δρόμο αυτό. Στις προτάσεις τη περασμένης εβδομάδας νομίζω ότι πραγματικά στερείστε της λογικής. θα πρέπει να γίνει αυτό το άλμα, αλλά θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια ισόρροπη πολιτική όπου θα συνδυάζουμε τη φορολογική υπευθυνότητα με ε, την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αφήσατε ορισμένε σημαντικέ επιλογέ που πράγματι θα οδηγούσαν σε αυτό το ποιοτικό άλμα στον τομέα. Πραγματική, πραγματικό συντονισμό τη οικονομική πολιτική θα πρέπει να οδηγήσει σε ε, περισσότερο διαφοροποιημένα ε, προγράμματα εξυγίανση αντί για αυτή την κοντόφθαλμη ατζέντα λιτότητα που δεν έχει καθόλου νόημα από οικονομική άποψη. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να, να, δημιουργηθούν ε, ε, θέσει απασχόληση από κοινού με τη φορολογική εξυγίανση. Σήμερα μειώνονται τα ελλείμματα, αλλά ει βάρο τη απασχόληση. Τρίτον, πρέπει να δούμε ε, και αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί σε επίπεδο ε, G20, συμπεριλαμβάνοντας ε, και τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών κτλ. Και ταυτόχρονα χρειαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις από εσάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε το, το, το, φορολογικό αυτό άχθος από την απασχόληση να αρθεί ως τον πιο γρήγορα, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένα κράτη-μέλη αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό. Και τέλος, ε, ε, αντί για αρνητικέ κυρώσει θα πρέπει να δείτε το θέμα των θετικών κινήτρων. Γιατί ε, ε, πραγματικά κάτι τέτοιο θα μα οδηγούσε σε μια αποτελεσματική πολιτική. Ελπίζω λοιπόν ε, να έρθετε στα λογικά σα και το φθινόπωρο να οδηγηθείτε σε μια πιο ισόρροπη δέσμη προτάσεων. Σα ευχαριστώ και τώρα να δώσουμε ε, το, το λόγο στον πρόεδρο Φερχόφστα εκ μέρου τη ομάδα των Φιλελευθέρων. Euh, Κύριε Πρόεδρε, είμαι ικανοποιημένο από την παρουσίαση του πακέτου από τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν μου επιτρέπετε να σε εκφράσω τη γνώμη μου, θα ήθελα να σας πω ε, να το καταθέσετε το συντομότερο δυνατό με βάση το δικαίωμα πρωτοβουλία σας. Το, ε, καταθέστε το στο τραπέζι του Συμβουλίου και στο τραπέζι του Κοινοβουλίου. Γιατί αυτή είναι η μηχανική και ο τρόπο λειτουργία τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν έχει την πρωτοβουλία. Καλή επιτυχία στην ε, ομάδα εργασία που δημιουργήθηκε, αλλά στην τελική φάση η Κομισιόν θα πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε τη και να καταθέσει μια πρόταση στο τραπέζι των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτό το πακέτο, Πρόεδρε, ε, παραμένουν κάποια ερωτηματικά. Το πρώτο και θεμελιώδες ερώτημα είναι ποιο θα διαχειριστεί αυτή την ε, διακυβέρνηση, την οικονομική διακυβέρνηση. Τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο ή τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σαφέ. Νομίζω ότι τα κοινοτικά θεσμικά όργανα θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Ποτέ δεν ε, ε λειτουργήσε ο αυτοέλεγχο από τα κράτη-μέλη. Ποτέ δεν λειτουργήσε στο παρελθόν και δεν πρόκειται να λειτουργήσει και στο μέλλον. Δεύτερον, κυρώσει ναι. Αλλά όχι μόνο κυρώσει ε, στο Σύμφωνο Σταθερότητα, γιατί όπω είπατε κι εσεί, είναι μία πτυχή τη πολιτική οι Θα πρέπει επίση ε, να ασχοληθούμε και με την ανταγωνιστικότητα ή και με τις διαφθορτικές μεταρρυθμίσεις ε, στις, στην ευρωπαϊκή οικονομία. Και εκεί πρέπει να προβλέψουμε κυρώσεις. Και εδώ θα ήθελα να ζητήσω να υποστούν τις ε, συνέπειες κάποια κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη λοιπόν απαιτούν κυρώσεις στο σύμφωνο σταθερότητας, αλλά όταν μιλάμε για κυρώσεις ε, στη στρατηγική 2020 για θέματα ανταγωνιστικότητας είναι πολύ πιο απρόθυμα. Ή το ένα ή το άλλο. Αν θέλουμε κυρώσεις, θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε σε όλους τους τομείς. Τρίτον, θα πρέπει επίσης, ε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να σκεφτείτε και μια στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε μόνο να πούμε ότι θα μειώσουμε τα ελλείμματα. Εντάξει, και εγώ είμαι παλιός ε, υπουργό Οικονομικών, μου αρέσουν τα ελλείμματα όταν μειώνονται. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να έχουμε και οικονομικές, ε, πολιτικές, πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης. Και ο μόνο φορέα που μπορεί να προωθήσει κάτι τέτοιο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορεί να δανειστεί, που έχει προγράμματα ε, υποδομών, πανευρωπαϊκών υποδομών. Τα χρειαζόμαστε. Ε, Όπω αναφέρονται στην έκθεση Μόντι. Με αυτόν τον τρόπο και η Κομισιόν μπορεί να κάνει προτάσει προ αυτήν την κατεύθυνση. Να μην μιλάτε μόνο για τη μείωση των ελλημάτων, που εντάξει χρειάζονται και αυτά, ε, σταθερότητα κλπ. Αλλά χρειαζόμαστε και μια αξιόπιστη στρατηγική οικονομική ανάπτυξη για να μην πέσουμε ε, στην παγίδα της, του οικονομικού τελματισ... Ε, αποτελμάτωσης όπως συνέβη στην Ιαπωνία τα τελευταία χρόνια. Επίσης, χαίρομαι για τη δημοσιοποίηση αυτών των αποφάσεων. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πριν από ένα χρόνο, όπως έκανε οι Αμερικανοί. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να τροφοδοτήσουμε την ιδιωτική πίστη και τελειώνω τέλο ε, τις μου με την οικονομική εποπτεία. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει συμφωνία με το Κοινοβούλιο εάν το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη δεν σεβαστούν ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή θα έχει το τελευταίο λόγο σε περίπτωση διαφωνία. Αυτό είναι το βασικό. Επίση υπάρχει και στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό. Αυτή ήταν η βάση τη της λογική. λογικής. Τα κράτη-μέλη όμω δεν το έχουν καταλάβει. Πρέπει να το καταλάβουν, Πρόεδρε. Και πρέπει να το δεχτούν. Αλλιώ θα υπάρξει συμφωνία για την εποπτεία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, κύριε Φερχόφσταντ. Πολύ, πάρα πολύ έμπλος ενθουσιασμού ο λόγος σας, αλλά είστε λίγο ε, μακροσκελής. Γι' αυτό σας διάκοψα. Ο κύριος Γκίγκολτ από τους Πράσινους έχει το λόγο. Ευχαριστώ για την παρουσίαση της ανακοίνωσης. Είναι σαφές νομίζω και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αγαπητοί συνάδελφοι εδώ. Ότι Υπάρχει ο κίνδυνος ε, σε μια τόσο δύσκολη κρίση που αντιμετωπίζουμε να επαναλάβουμε τα παλαιά πρότυπα, δηλαδή τα δημοσιονομικά ελλείμματα, να τα συνδυάσουμε με τα, με τα προβλήματα και τα ελλείμματα στην ανταγωνιστικότητα. Η επιλογή της λιτότητας δεν μπορεί να μας ε, βοηθήσει να προχωρήσουμε και γι' αυτό θα πρέπει με την πρόταση που βλέπουμε να διαπιστώσουμε ότι περιλαμβάνονται και σημαντικές πρόοδοι, σημαντικές πρόοδοι όσον αφορά το συντονισμό των προϋπολογισμών, δηλαδή του δημοσιονομικού σχεδιασμού και εκεί όπου υπάρχουν σαφώς ε, ανισορροπίες που μέχρι τώρα δεν υπήρχε δυνατότητα καν να συζητήσουμε με σοβαρότητα για τέτοια ζητήματα, για και ε, ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, τώρα ήρθε η στιγμή να συστήσουμε ακόμη και για κυρώσεις. Πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε. Έχει έρθει η στιγμή, ο πολίτης δεν ανέχεται περαιτέρω ε, να συνεχίζεται αυτή η κρίση, να υπάρχουν φορολογική παράδειση, να υπάρχουν ε, μεγάλα τμήματα της δημόσιας οικονομίας, των δημόσιων οικονομικών που ε, εκφεύγουν τη φορολογία. και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες εξηγήσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Η δημοσιονομική πολιτική όμως δεν αρκεί να, να συντονίζεται κατά τον τρόπο με τον οποίο μας τον περιγράψετε. Πρέπει δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να δράσει και αντικυκλικά, πράγμα το οποίο όμως δεν βλέπω μέσα στο κείμενό σας. Και παραμένει από ό,τι φαίνεται ταμπού το να λέμε ότι σε περίπτωση μίσους και λυσμένων προϋπολογισμών ε, υπάρχουν ε, αυτά τα χαρακτηριστικά σε ορισμένα κράτη ε, τα οποία έχουν υψηλό χρέος, τα οποία έχουν μεγάλα ελλείμματα και ίσως θα πρέπει αυτά να τα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα, όπως πρέπει να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα και τα προβλήματα των της φούσκας που εμφανίζεται σε ορισμένες αγορές. Γι' αυτό παρακαλούμε να κοιτάξουμε όλες τις παραμέτρους της κρίσεως. Ας μην προσπαθήσουμε μόνο να δώσουμε λύσεις στα βιαστικά. Ο πολίτης της Ελλάδας περιμένει, της Ευρώπης να περιμένει μια γενική λύση που θα φύγει όλα τα κακό σκήμενα. Ευχαριστώ κυρία Σουίνμπερν από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Κυρία Σουήπον. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα ε, τα οποία ε, σχετίζονται με την οικονομική κρίση και θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε ε, να υιοθετήσουμε μια ισχυρή και ανθεκτική δομή ώστε το πιο γρήγορα. Έτσι ώστε να υπάρξει ένα κοινό σύνολο κανόνων. Έτσι ώστε να αναλάβουν τι ευθύνε του και τα κράτη-μέλη σε επίπεδο οικονομική διακυβέρνηση αλλά και σε επίπεδο χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια συνένεση και το αποτέλεσμα πρέπει να εφαρμοστεί αυστηρά και από τα 27 κράτη-μέλη και να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση. Όλα, ε, ε, και θα πρέπει ε, αυτοί οι φορεί να φροντίσουν έτσι ώστε να στρατολογήσουν και να προσλάβουν το κατάλληλο προσωπικό. Πρέπει να δώσουμε ένα σαφέ μήνυμα ότι όλε αυτέ οι διαδικασίε και οι υποπτικέ αρχέ, ιδιαίτερα όσον αφορά το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, ότι αυτέ οι αρχέ λοιπόν είναι απαραίτητε και θα, και θα λειτουργήσουν ει όφελο των πολιτών. Η πρόσφατη οικονομική κρίση οδηγεί στην ανάγκη για λήψη αυστηρών και σημαντικών μέτρων θα πρέπει να μειώσουμε τι διαφορέ ανάμεσα στι αγορέ, να βελτιώσουμε τη διαφάνεια ε, στο σύνολο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ε, η πρόσφατη συμφωνία θεωρήθηκε ε, ότι ε, θέτουμε τη μεταρρύθμιση στο δομέα αυτό ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αν συμφωνήσουμε στις προσεχείς ημέρες τότε θα έχουμε ένα σημαντικό πλαίσιο και έτσι ώστε και οι τρεις επιτροπές Λαμφαλούση να γίνουν ευρωπαϊκές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του και με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί και η λειτουργία λειτουργία τη εσωτερική αγορά στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όμω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε νέα αρχή ε, θα ε, λειτουργεί ε, σε συντονισμό με, με, τους, με εθνικούς φορείς και οι διαπραγματεύσεις πάντα θα πρέπει να οδηγήσουν στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Το θέμα δεν είναι κατά πόσο θα έχουμε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη. Πραγματικά πιστεύω ότι ακολουθεί τη σωστή οπτική γωνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι, τελικά θα καταλήξουμε σε ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα σύστημα το οποίο θα είναι προ όφελο των οικονομιών μα γενικά. Σα ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει ο κύριο Μπίσκι από την Ενωμένη ΕΕ. Αριστερά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι τελευταίε ε, εβδομάδε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφερε ομπρέλα ασπίδα προστασία για το ευρώ και τη μεγάλη στρατηγία για το 2020. Φαίνεται όμως ότι προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε το ότι αφενός μεν έχει διασώσει τις τράπεζες αφετέρου δεν προχωρήσει από διάρθρωση των κοινωνικών συστημάτων και των συστημάτων ασφάλισης. Αυτέ οι προτάσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης κατά την άποψή μα προχωρούν προς την εσφαλμένη κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως άλλωστε ήδη στη, προέκυψε από την ομάδα εργασία υπό τον πρόεδρο του Συμβουλίου Φαν Ρομπόι, να τροποποιήσει όχι κατά το περιεχόμενό του το σύμφωνο, αλλά να ενισχύσει μόνο τι κυρώσει και να επιβάλλει μέτρα για τα κράτη που παρουσιάζουν έλλειμμα, όπω άλλωστε θέλει και το Συμβούλιο. Πράγμα το όμω το οποίο δεν έχει φέρει αποτελέσματα στο παρελθόν, ούτε και πρόκειται και στο μέλλον να φέρει αποτελέσματα. Το Κοινοβούλιο πάντω εκφράσει την ικανοποίησή του τουλάχιστον οι χειρότερε προτάσει περί κρίσεων για τα κράτη που παρουσιάζουν έλλειμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έγιναν δεκτέ. Η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι αδύρυτο η ανάγκη. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή ε, προσπάθεια να αποπληρωθεί το χρέος και πλέον πρέπει το ε, Συμβούλιο να ανασκουμποθεί. Δεν πρόκειται να δώσουμε λύση αν προσπαθήσουμε να μειώσουμε το εθνικό έλλειμμα σε σε επίπεδο 3% μέσα σε ένα χρόνο για να φτάσουμε στους στόχους του Μάστριχτ. Αυτό μόνο σε νέο χρέος μπορεί να οδηγήσει. Οι ανισορροπίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αρθρωτικές ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν γιατί αυτές είναι ακριβώς που εκμεταλλεύονται οι κερδοσκόποι. Έτσι λοιπόν τα ε, επιτυχημένα, τα ισχυρά κράτη θα πρέπει να σταματήσουν την επιθετική τους ε, συμπεριφορά απέναντι στα άλλα, στα λιγότερο ισχυρά. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να ενισχυθούν οι εσωτερικές αγορές και η, η ζήτηση στα ασθενέστερα οικονομικά κράτη. Δεν χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση των κυρώσεων, αλλά εκ των βάθρων αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Κύριο Μπλουμ από την Ευρώπη τη Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπη. Στην τελευταία σύνοδο, κύριε Πρόεδρε, ε, φύγατε νωρί και χάσατε τα λόγια σοφίας μου. Ελπίζω σήμερα να μπορέσω να προσφέρω κάποια άλλα λόγια σοφίας. Τι να σα πω. Ε, σας λυπάμαι πραγματικά, αλλά φταίτε κιόλα. Με το σημερινό οικονομικό πείραμα, είναι πείραμα, το οποίο νομίζω θα αποτύχει. Θυμάμαι μία ε, ομιλία που άκουσα στην δεκαετία του 90 στο Cambridge ε, που εξηγούσε γιατί θα αποτύχανε. Και τώρα, δέκα χρόνια μετά, φαίνεται ότι μάλλον δίκιο είχανε. Και με το εγχειρίδιό σας ε, πάλι απεδείχθη λάθος. τελικά εσείς όμως το σκίσατε αυτό το εγχειρίδιο ε, οποιαδήποτε δυσλειτουργική οικονομία ε, τη δεχτήκατε στην Ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ε, με αυτόν τον τρόπο επιταχύνατε το θάνατο της Ευρωζώνης. Δεν θα πρέπει να σας εκπλήσει λοιπόν που θα πεθάνει το ευρώ. Αυτό ήταν προαναγγελθής θάνατος. Και τώρα, εγώ θυμάμαι ότι αγόραζα ε, ευρωμόλογα, αγόραζα ομόλογα στο City ελληνικά. Νομίζω ότι οι εμπορικές τραπεζές μας αντιμετώπισαν τροπέρα, τρομερά προβλήματα. Στην πραγματικότητα αγόρασαν αυτά τα, αυτούς τους τίτλους, τους αναπακετάρισαν και τους ξαναπούλησαν ε, με χασούρα. Αγοράζουν ε, σκουπίδια ομόλογα ε, τα πουλάνε και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το χάλι. Αν θέλετε να φύγουμε από αυτό το χάλι θα πρέπει νομίζω να ξεφορτωθείτε αυτό το πολιτικό α, κατεστηγμένο το οποίο υποστηρίζει τις τράπεζες. Ε, γιατί είναι τμήμα του προβλήματος και όχι της λύσης. Madame... Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρίν Λεπέν. Αυτή τη στιγμή η ζώνη του ευρώ ε, βρίσκεται μπροστά σε μια οικονομική ιστορία, ε, κρίση, ε, την, πρώτη, την πιο σημαντική στην ιστορία της. Μείωση ανταγωνιστικότητας, μείωση επασχόλησης κτλ. Και αυτό το είδαμε πρόσφατα και με την κρίση στην Ελλάδα και με την κρίση που σύντομα θα φτάσει στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Άρα γενικευμένη φτώχεια των πολιτών στις χώρες αυτές. Μιλήσατε για οικονομική σύγκληση, υποσχεθήκατε τη σύγκληση. Σήμερα όμως μας οδηγείτε στη χρεοκοπία. Ε, εσείς έχετε την ευθύνη αυτής της ε, τραγωδίας, διότι επιβάλλοντας μια ενιαία, ομοιόμορφη και απολυταρχική νομισματική πολιτική σε τόσα διαφορετικές οικονομίες, ευνοείται την κερδοσκοπία. Ε, και, την οικονομική κρίση. Ε, το 2007 είχε οικονομικό πλεόνασμα ε, η Ισπανία και σήμερα ε, ε, βρίσκεται μπροστά σε ένα έλλειμμα 12%. Γιατί, γιατί το ενιαίο νόμισμα οδήγησε σε μια τρομερή κερδοσκοπία στι τιμέ των ακινήτων και σήμερα αυτή η χώρα είναι γεμάτη άδεια σπίτια. αυτή η νέα κρίση με τα subprime είναι γενικευμένη και μεταδίδεται πολύ γρήγορα. Και συνεχίζεται όμω συνεχίζεται αυτή τη λανθασμένη πολιτική ε, ε, μιλώντας, μιλώντας για ενιαίο έλεγχο ε, και επιβάλλοντας στους πολίτες της Ευρώπης μια πολιτική λιτότητας χωρίς προηγούμενο. Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για να κάνετε τις τελευταίες παρατηρήσεις. Σα ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιε ε, συγκεκριμένε ερωτήσει που έγιναν. Πρώτα απ' όλα στην κυρία Μάρτιν Κόλ, σα ευχαριστώ για την υποστήριξή σα. Πράγματι πιστεύουμε ότι ε, με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η αξιοπιστία του Συμφώνου Ανάπτυξη και Σταθερότητα αλλά και του ευρώ ε, και του ευρωπαϊκού σχεδίου στο σύνολό του. Και αυτό βεβαίω ε, θα γίνει με ε, όλε αυτέ τι προσπάθειε από κοινού. Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που ε, παρευρεθήκε και ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπαμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται για όλες για την πρόοδο των συζητήσεων όσον αφορά τη μελλοντική οικονομική διακυβέρνηση τη Ευρώπη. Ορισμένε από τι ανησυχίε που εκφράστηκαν από τον κύριο Χιού και από τον κύριο Μπίσκι. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να εξεταστούν με προσοχή. Αλλά νομίζω ότι η πρότασή μα ε, ακριβώ αυτό κάνει. Λαμβάνει υπόψη τι ανησυχίε σα. Γιατί εσεί λέτε ότι ε, το, το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη δεν ε, αποτελεί πανάκια. Και συνδέουμε την ανάλυση τη εφαρμογή των μέτρων σταθερότητα στα πλαίσια του συμφώνου με ε, τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και με τα προβλήματα ε, σύγκλησης, απόκλησης μάλλον. Άρα λοιπόν ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση που δεν αφορά μόνο τη μακροοικονομική συνιστόσα, αλλά και την ανάπτυξη, όπως ακριβώς είπε και ο Κίβερ Χόφστατ, που εξετάζει και την καινοτομία και τις μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Μα αυτός είναι και ο στόχος μας, από κοινού με την, με, την ομάδα G20. Και ακριβώς τώρα μας απασχολεί και το θέμα της ιστορικής αγοράς. Και με βάση την έκθεση του Μάριο Μόντι έκθεση που του ζητήσαμε να υποβάλει. Τώρα ε, καταβάλουμε προσπάθεια και θα έρθει και ο κύριο Μπαρνιέ ε, το φθινόπωρο με πολύ σημαντικέ ε, προτάσει ε, στα πλαίσια τη ιστορική αγορά, ακριβώ για να δούμε τα προβλήματα αυτά. Η πρότασή μα λοιπόν δεν αφορά ε, μόνο ε, τον προληπτικό έλεγχο σε μακροοικονομικό επίπεδο, αλλά σήμερα το θέμα μα είναι η οικονομική διακυβέρνηση. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι ακριβώ δεν πήγε καλά. Το τονίζω. Όμω εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τη μακροοικονομική συνιστόσα και την ε, προφύλαξη αλλά ε, και με την οικονομική ανάπτυξη. Και βεβαίως σε τελευταία ανάλυση ε, θα συμφωνήσουμε το σχέδιο αυτό, αλλά για πρώτη φορά έχουμε μια συνολική, μια ολιστική προσέγγιση, προσπαθώντα να εξετάσουμε όλε τι πτυχέ. Θα θυμάστε ότι πριν από λίγου μήνε, όταν ε, ε, παρουσίασε στρατηγική για την Ευρώπη 2020, ορισμένοι είπαν ότι όχι, δεν μπορείτε να τη συνδέετε με το σύμφωνο ανάπτυξη θερότητα, γιατί μπορεί να αποδυναμώσει το σύμφωνο. Τώρα όλοι όμω συμφωνούν στο ότι πράγματι θα πρέπει να συζητήσουμε του μακροοικονομικού περιορισμού ε, και δεν έχει νόημα να συζητάμε του μακροοικονομικού περιορισμού ε, χωρί να εξετάζουμε ε, τι μεταρρυθμίσει, την ανάπτυξη, την απασχόληση. Ακριβώ και στα πλαίσια τη Ευρώπη 2020 μιλούσαμε για, τους, για τη μείωση των παραγόντων αποκλεισμού, εκπαίδευση, απασχόληση κτλ. Άρα λοιπόν εδώ προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε όλα τα μέσα τη οικονομική πολιτική, να, να δούμε και την ευρωπαϊκή διάσταση και την εθνική διάσταση και ταυτόχρονα έχουμε στόχου που αφορούν την ανταγωνιστικότητα την ε, κοινωνική ένταξη και την εκπαίδευση. Έχετε δίκιο κύριε Φερχόφστατ. Η Κομισιόν πρέπει να κάνει τις προτάσεις. Αυτό κάνουμε. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση αυτή η σημερινή. Γι' αυτό ακριβώς όλοι ρεν συνεισφέρει και αυτός ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Task Force. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω να υπάρξει συνένεση γιατί Αυτές είναι πολύ σημαντικές αλλαγές. Φυσικά, κάποια στιγμή θα πρέπει να παρουσιάσουμε τι συγκεκριμένε νομοθετικέ προτάσει ω Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ε, σε αυτή την προσπάθεια να εμπλέξουμε και το Κοινοβούλιο. Επίση, σε αυτή την ε, συνολική προσέγγιση να έχουμε και μακροοικονομική εποπτεία. Δεν μιλάμε μόνο για κυρώσει, για εκείνου που δεν ε, πληρούν τα κριτήρια για το χρέο και τα ελλείμματα. Θα προσπαθήσουμε επίσης να ενδυναμώσουμε τον συντονισμό σε ό,τι αφορά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες όπου αυτές υπάρχουν. Επίσης αναφέρατε, ορισμένοι από εσά, ορισμένα πράγματα. Από το 2011 μια και η δική μας μεταρρύθμιση βασίζεται σε τη νέα δομή, χρειαζόμαστε όλα τα στοιχεία. Τις τελευταίες μέρες η νέα Βελγική Προεδρία έχει δώσει νέα ορμή. Και οι δύο πλευρές νομίζω ότι δείχνουν ρεαλισμό. Ε, χαίρομαι για τη φιλοδοξία που δείχνει το Κοινοβούλιο ε, και χαίρομαι για την στεναρή υποστήριξη που μας δείχνει. Θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνετε ό,τι μπορείτε, ούτως ώστε να υπάρξει τις επόμενες μέρες μια ικανοποιητική α, συμφωνία. Νομίζω ότι Είμαστε πολύ κοντά. Με διάφορα συμβαστικά κείμενα η Κομισιόν έχει συνεισφέρει και με μεγάλη χαρά σημειώνει την πρόοδο που βλέπει και θέλουμε τώρα οι δύο σύνομοθέτες να διατηρήσουν αυτό το δυναμικό. Όπως είπε η κυρία Στρίνμπερν, και έχει πολύ σωστά, οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν την πολιτική συμφωνία, αλλά δεν έχουν ακόμα την νομοθεσία. Όταν διαβάζετε τις εφημερίδες, ε, μας δίνει την εντύπωση ότι οι Αμερικανοί είναι πολύ πιο μπροστά από εμά αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Ο πρόεδρος Ομπάμα στο G20 είπε ότι Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των μερών. Μπράβο. Αλλά εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε την νομοθετική μας προσπάθεια πολύ πριν τους Αμερικανούς και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε και τον ηγετικό μας ρόλο ε, στην ε, χρηματοπιστωτική εποπτεία και ρύθμιση και να διατρανώσουμε το ρόλο της Ευρώπης ε, στον τομέα αυτό. Ορισμένοι από εσά μιλήσατε για τα τεστ αντοχής. Η Κομισιόν προωθεί την ε, διαφάνεια και κοινοποιεί τα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων αυτών ε, τεστ αντοχής των ε, τραπεζών. Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησαν να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα, αλλά είμαι πραγματικά ικανοποιημένο με τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να γίνει κάτι πιο. Να υπάρχει δημοσίευση. Με αυτόν τον τρόπο θα καθησυχάσουμε του επενδυτέ είτε θα... και θα άρουμε τι αβάσιμε ανησυχίε και θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ακόμα υπάρχουν. Είμαι πεπισμένο ότι η αντοχή των ευρωπαϊκών τραπεζών και του ευρωπαϊκού ε, τραπεζικού συστήματο θα αποδειχθεί, αλλά θα πρέπει να δούμε του θύλακε ε, ε, τη αδυναμία και του ευάλωτου θύλακε και να του αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να έχουμε μηχανισμού για να του ενεργοποιήσουμε σε περίπτωση που χρειαστεί και ακόμα μια φορά αυτό είναι εθνική ευθύνη. Ε, αν χρειαστεί κρατική παρέμβαση, θα εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαίρως ε, με βάση τους κανόνες ε, για τις κρατικές ενισχύσεις. Η ευρωπαϊκή απόφαση ελήφθη με πολύ θετικό τρόπο από το G20 στο Τορόντο για να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα των τεστ αντοχή. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο τρόπο για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο συνολικό μα ε, ευρωπαϊκό σύστημα. Όπως βλέπετε, αγαπητοί βουλευτές, βρούμε σε πολλαπλά μέτωπα. Σήμερα σας παρουσίασα τις προτάσεις τις πιο πρόσφατες ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Αλλά δεν θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις προτάσεις αυτές από τις άλλες προσπάθειες, παράλληλες προσπάθειες που κάνουμε ε, για να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην οικονομική μας πολιτική ε, για να καταλάβουμε ότι η ΟΝΕ ναι, χωρίς κάποιο οικονομικό συντονισμό δεν έχει κανένα νόημα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον όλων των πολιτών ε, προς τη σταθερότητα του ευρώ. Ε, είναι καλό βέβαια για την Ευρωζώνη, αλλά νομίζω ότι είναι καλό για όλη την Ευρώπη. Και όλων όσων θέλουν ανοιχτές αγορές, ανοιχτές οικονομίες και ανοιχτές κοινωνίες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την προσέγγιση και για την ε, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ολοκληρώνει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Και τώρα, με βάση τη μερίσια διάταξη, θα κάνω μια κοινή